Okay. Hanu, there's a place for you. <laughs> so, guten Morgen. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής ε, στην ε, τρέχουσα θητεία. Υποθέτω ότι όλοι σας είσαστε κάπως λυπημένοι. Λίγο, λίγο, εν πάση περιπτώσει. Ε, να σας ρωτήσω αν ε, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Το σημείο 7 θεωρώ ότι δεν το χρειαζόμαστε πλέον, δεν χρειάζεται συνεδρίαση των συντονιστών, γι' αυτό λοιπόν το ε, σημείο 7 διαγράφεται. Και περνάμε στο δεύτερο σημείο τη ημερήσια διάταξη, έγκριση των πρακτικών, Ως συνήθω τα πρακτικά τη τελευταία συνεδρίαση της 18 Μαρτίου είναι στη διάθεσή σα. Αν δεν ακούσω ενστάσει κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση, θεωρώ ότι είναι εγκεκριμένα. Δεν έχουμε βουλγαρικά, σλοβένικα ή κάποιες άλλες γλώσσες. Τα ελληνικά πάντως μπορείτε να τα μιλάτε και να τα ακούτε χωρίς πρόβλημα. Βρίσκεται λοιπόν ε, και μία έκθεση για την ε, αποστολή στη Ρήγα. Εγώ προσωπικά να σας συστήσω να πάτε στη Ρήγα. Είναι και πολιτισμική πρωτεύουσα φέτος. Είναι πραγματικά μία πόλη της μουσικής μια εκπληκτική πόλη με Jugendstil. Αυτό δεν το γνώριζα. Αν θέλετε λοιπόν το καλοκαίρι να κάνετε ένα ωραίο ταξιδάκι στη Βαλτική, να πάτε και θα χαρούν και πολύ να σας δουν γιατί η απειλή από την Ανατολή είναι κάτι το οποίο υφίσταται, είναι πραγματικό και πάντα χαίρονται λοιπόν τα κράτη αυτά όταν βλέπουν επισκέπτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αξιαγάπητα τα κράτη αυτά. Στο τέσσερα λοιπόν τώρα τη ημερήσιας διάταξη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους. Μία παλιά οδηγία που χρήζει ανανέωσης. Και η κυρία Βερζιά ήταν ε, ε, αρκετά ευγενική για να λάβει την ε, έκθεση αυτή. Ξέρετε ότι δεν ήταν εύκολο αυτό, γιατί είναι δύσκολο το νομικό αυτό εγχείρημα και δεν έχουμε και τόσο πολλούς νομικούς εδώ στην Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνέβαλε. Κυρία Βεριά, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσοι εργάστηκαν πάνω στο θέμα. Είναι ένας φάκελος πολύ τεχνικός και ιδιαίτερα ε, με νομικά ζήτημα. Κάναμε μια εξαιρετική εργασία. Ευχαριστώ επίσης και την Πρόεδρο σας, ε, δηλαδή, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες. Το Κοινοβούλιο εξήλθε με το κεφάλι ψηλά σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Ευχαριστώ κυρία Δεργία. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Έχουμε μία και μόνο ψηφοφορία. Να σας παρακαλέσω λοιπόν να ψηφίσετε έναρξη της ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας. Όχι. 10... Α, συγγνώμη, να ξαναξεκινήσει η, η συνεδρίαση. Τώρα λοιπόν ένοιξε η συνεδρίαση. Κυρία Παλιαδέλη. The vote is closed. Πέρασε τις ψηφορίες. It 13. 13, λοιπόν, η ψήφη υπέρ. 14 have voted, 13 14 ψήφοι, 13 υπέρ, 1 κατά. We check, we check if you have voted. We are 14. Ναι, μα κοιτάξτε, μία και μόνο ψηφοφορία έχουμε. Πόσο λάθος μπορεί να πάει. Άλλη μια φορά. Άντε, μην το επαναλάβουμε. Ναι, ναι, τώρα όχι, δεν γίνεται τίποτα. σα παρακαλώ. Μόνο για τον Σαντιάγκο, γιατί θέλω την προσοχή μας σήμερα. Α ψηφίσουμε λοιπόν άλλη μια φορά έναρξη τη ψηφοφορίας. Ωραία. 14 ψήφοι. Υπέρ, 14 ε, υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Βερζιά, ήταν δύσκολο το έργο σας. Και τώρα να περάσουμε στο 5 τη ημερήσιας διάταξη για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Χαίρομαι που δεν αναγκαστήκαν όλοι να παραστούν στον τριμερή διάλογο, γιατί ήταν πραγματικά δύσκολο το εγχείρημα το Συμβούλιο. Ήταν πολύ ε, αμετακίνητο. Και δεν ήθελε να πούμε ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες χρειάζεται μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό ειλικρινά ποιος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, πολιτιστική πρωτεύουσα και το Συμβούλιο θέλει να βγει η λέξη ε, Ευρωπαϊκή Διάσταση. Αναρωτιόμαστε λοιπόν σε ποιο πλανήτη ζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το συζητήσαμε λοιπόν επί μακρόν και καταφέραμε να το πετύχουμε αυτό και επίσης καταφέραμε αυτή η επίπονη διαδικασία κάπως να αποδυναμωθεί. Ξέρετε, όταν, ορίζεται, όταν οριζόταν η πολιτιστική πρωτεύουσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι εμπειρογνώμονε το ανακοίνωναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εμά, στο Συμβούλιο. Έπρεπε να το συζητήσουμε, να το ψηφίσουμε. Μόνο ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ποιο θα έλεγε, ποιο θα τολμούσε να πει όχι προ ε, την απόφαση ενό πάνελ εμπειρογνώμων. Εμεί λοιπόν λέγαμε ναι, συμφωνούσαμε, συμφωνούσε και το Συμβούλιο. Ανακοινωνόταν τότε λοιπόν η πρωτεύουσα έξι μήνε τουλάχιστον. Για το τίποτα δηλαδή. Και γι' αυτό λοιπόν χαρήκαμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη διαδικασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει μετά την απόφαση του πάνελ την ε, πρωτεύουσα. Το Συμβούλιο όμως δεν συμφώνησε. Τρεις φορές, τρεις φορές αναγκαστήκαμε να διαβουλευτούμε με το Συμβούλιο μόνο για το θέμα αυτό. Έλεγε το Συμβούλιο, μα όχι, το Συμβούλιο πρέπει να κάνει την ανακοίνωση και το Συμβούλιο δεν είναι και τα λεφτά. Και είπαμε στο Συμβούλιο ότι κοιτάξτε, δεν δίνεται και τίποτα ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο. Σύμφωνοι, αλλά τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά είναι από τον κοινό προϋπολογισμό. Και μόνο η χώρα ε, που ε, έχει την πρωτεύουσα μπορεί να το ορίσει αυτό και καταφέραμε, εν πάση περιπτώσει, να το πετύχουμε, αλλά ώρες μας πήρε, ώρες ε, συζητήσεων. Χαίρομαι που αυτά τα ακούν οι πολίτες. Πόσο αμετακίνητο και, τι να πω, ε, συμβούλιο του σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε κι άλλο ένα πρόβλημα, δεν ήθελαν να μπει το urban planning, urban development, η αστική ανάπτυξη. Εμείς ε, υποστηρίξαμε το εξή, ότι αν υπάρχει μια πολιτιστική πρωτεύουσα θα πρέπει να φροντίσουμε η δραστηριότητα να έχει να κάνει και κάτι με την ε, χωροταξία, την αστική, με τον πολιτισμό κτλ. Ούτε αυτό το ήθελαμε, το καταφέραμε παρόλα αυτά να μπει. Τα πετύχαμε λοιπόν όσα θέλαμε, ε, αλλά μας πήρε χρόνο. Τρεις προεδρίες περάσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι καλό πλέον. Και τώρα λοιπόν καλούμαστε να ψηφίσουμε γι' αυτό λοιπόν. Α, συγγνώμη, δεν ξέρω, θέλει κάποιο να πάρει το λόγο. Κανεί, τίποτα. Ωραία. Άρα, έναρξη τη ψηφοφορία. Πέρα. 15 ψήφοι. Υπέρ. 0 αποχές, 0 ψήφοι κατά. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ποιος ήταν υπεύθυνο? Α, ο Ιβαν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τη δουλειά σας. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει μέσα στα διάφορα. Στο 6 θα ήθελα να σας ανακοινώσω το εξή. Στην τελευταία περίοδο κοιτάξαμε το θέμα της ευρωπαϊκής ε, ε, σφραγίδας, ε, πολιτισμικής σφραγίδας. Μήπως την ηγεσία της κυρίας Παλιαδέλη. Και τη Δευτέρα Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε λοιπόν την πρώτη τέτοια αυτή πλακέτα για την πολιτισμική κληρονομιά Καρτάνου ανασκαφή ρωμαϊκή με πολλά ε, εκπαιδευτικά στοιχεία, πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σημαντική. Και μετά, λοιπόν, στη Χάγη Έχουμε τον ε, οίκο των παλάτι της Ειρήνης στο Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο με μακρά ιστορία και εκτός αυτού έχουμε και ένα στρατόπεδο ναζί στη Χάγη στο οποίο επισκέφτονται πάρα πολλά σχολεία κάθε χρόνο Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό το μείγμα. Το τρίτο, κύριε Παλιαδέλη, ποιο ήτανε. I do not remember. Α, Ρίγα. Ναι. Στη Ρίγα. Όχι, στο Ταλίν, στο Ταλίν, στο Ταλίν, ναι. Ένα εξαιρετικό μουσείο. Το μουσείο των συντεχνιών. Πολύ σημαντικό και στην Βόρεια Γερμανία και στη Ρίγα και στο Ταλίν μοντέρνα τεχνολογία προκειμένου ο κόσμος που επισκέπτεται το μουσείο να ενημερώνεται για την ιστορία μέχρι τον Μεσαίωνα. Έχουν λοιπόν αυτή τη σφραγίδα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αυτά λοιπόν υπενθυμίζουν την κοινή μας ιστορία. Αυτό είναι ο σκοπό, να υπενθυμίζουν ε, στο κοινό την κοινή μα ιστορία. Κάτι άλλο να πω ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε να με διορίσει για συντονίστρια για το βραβείο Λουξ. Για τον απλό λόγο ότι ενδεχομένως να εξαφανιζόταν το βραβείο αυτό αν δεν δαπανούσαμε τον απαραίτητο χρόνο. Και νομίζω ότι προτού γίνω πρόεδρος, αυτή η... αυτό το βραβείο δεν έπαιζε και δίτερο ρόλο εδώ στην Επιτροπή μας, γιατί ήταν πράγματα που τα μαθαίναμε από τις ανακοινώσεις. Γι' αυτό λοιπόν όταν μου ζήτησαν να αναλάβω αυτό το συντονισμό, είπα ότι ήθελα να το κάνω. Όχι για να τιμηθώ εγώ, αλλά για να προωθήσουμε και στους νέους βουλευτές αυτή τη νέα, αυτή την ιδέα του βραβείου Λουξ, για να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο επικοινωνίας. Και γι' αυτό λοιπόν χάρηκα ιδιαίτερα και σίγουρα θα το ξαναπούμε. Νομίζω ότι από κοινού πρέπει να εκτελέσουμε αυτό το καθήκον, αυτό το έργο. Και μια και είναι και η τελευταία συνεδρίαση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τη γραμματεία μας. Για να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες που περιτρίγησαν τον Στίβεν από εδώ. Δέκα γυναίκες νομίζω περιτριγύρισαν. Ιδιαίτερα ευγνώμονες είμαστε για την συνεργασία, πραγματικά υψηλή ποιότητα συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και θα ήθελα να υπογραμμίσω δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι έτσι σε όλες τις επιτροπές, αλλά εδώ σε αυτή την επιτροπή μου έκανε εντύπωση το πόσο καλή ήταν η συνεργασία. Δεν ήθελα, δεν θέλω να του αναφέρω όλου ονομαστικά, αλλά και τον επικεφαλής της γραμματείας Ασφαλώ να ευχαριστήσω και ελπίζω τον ε, επόμενο καιρό να έχετε εξίσου καλούς συναδέλφους, έναν ή μία καλή, καλό πρόεδρο που να εκτιμά και τη συνεργασία σας και κατακάσατε πιθανότητα και έναν ε, καινούργιο επικεφαλή στη γραμματεία, γιατί ξέρετε έχουμε και κινητικότητα στο Κοινοβούλιο που φροντίζει να, αλλάζουμε θέσεις, ε, να αλλάζουν θέσεις οι υπάλληλοι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους Κάποιοι είναι εδώ, κάποιοι είχαν αντικατασταθεί γιατί δεν ε, μπόρεσαν να είναι εδώ πέρα σήμερα. Έχει ξεκινήσει και η προεκλογική εκστρατεία. Να ευχαριστήσω όλου όσοι συνεργάστηκαν και εργάστηκαν και η επιτροπή αυτή ουσιαστικά ήταν ε, μια επιτροπή ξεχωριστή εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί πραγματευόμαστε, ξέρετε, θέματα τα οποία δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενα. Ναι, εντάξει, σε κάποιε περιπτώσει, κυρία Βερζιά, ήταν τα θέματα αυτά αμφιλεγόμενα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το Erasmus Plus κτλ. Ξέρω ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι όλοι είμαστε, έχουμε μια υψηλή πολιτισμική ε, ανάπτυξη. Όλους μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση, η κατάρτιση, το μέλλον των παιδιών μας, τη επόμενης γενιάς και θεωρώ λοιπόν ότι ήταν εξαιρετικά η συνεργασία και δεν έχουμε τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν, αν θέλετε, νομοτελειακά τις υπόλοιπες επιτροπές, γιατί έχουν και ιδεολογικό πώς άλλες διαφορές. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία και την ευτυχία να έχουμε μια καλή συνεργασία και θα ήθελα λοιπόν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τη συναδελφικότητά σας. Νομίζω ότι η συνεργασία ήταν και, και ευχάριστη σε πολλές περιπτώσεις μας. Ε, γέμισε χαρά. Και τα πολλά ταξίδια που έκαναν πολλοί εξημών μας έφεραν και πιο κοντά, αν θέλετε, στα πλαίσια της εργασίας της Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό και σε βάθος χρόνου θα αποφέρει, ξέρετε, καρπούς και πολιτικές φιλίες. Ξέρετε, οι πολιτικές φιλίες είναι κάτι δύσκολο να διατηρηθεί, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα το πετύχουμε. Γιατί πολλοί από εμά συζητήσαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν μόνο, ξέρετε, θέματα της Επιτροπής μας και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι χάσαμε και έναν συνάδελφο, έναν αξιότιμο και άξιο συνάδελφο, συνάδελφο όλοι μας άξιοι, Λούτα Μπίσκι, αναπληρωτής μου. Και ξέρω λοιπόν ε, ότι όλοι τον εκτιμούσαμε και ήθελα να τον αναφέρω στην τελευταία συνεδρίαση. Τι να σας πω, μου φαίνεται δύσκολο τώρα που σας ε, αποχαιρετώ, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Σας εύχομαι και μας εύχομαι στο μέλλον να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία και να υποστηρίζουμε που και που και το βραβείο Λουξ. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ είμαι κάπως συγκινημένη, ξέρετε, είναι και η τελευταία συνεδρίαση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό εξ ονόμαστος όλων των συναδέλφων και να επευθύνω και τις ευχαριστίες μου προς την Πρόεδρο. Νομίζω ότι όλοι εδώ θα αισθανθούμε την έλλειψη της εξαιρετικής σου Προεδρίας. Ήσουν πάντα πολύ ε, τηρούσε τα χρονικά όρια, ξεκινούσες πάντα στην ώρα σου, ανοιχτά μιλούσες, ποτέ δεν ε, κατέφυγες σε επεκφυγές ούτε μπροστά σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή λοιπόν ε, αυτή η διάθεση να μιλάς ανοιχτά είναι κάτι που θα μας λείψεις και νομίζω λοιπόν ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ε, πρέπει να σε ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έκανες. Σας ευχαριστούμε. Uh, και εγώ πρόεδρε. Θα σας αποχαιρετήσω, θα μιλήσω φιλανδικά γιατί είναι πιο εύκολο για μένα. Αλλά πάντα είμαι σύντομος όπως ξέρετε. Θέλω λοιπόν και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά που κάναμε μαζί. Νομίζω ότι είσαι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, γνωρίζεις πολύ καλά τα θέματα και σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια. Θα μας λείψεις. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να ξαναειδωθούμε κάποτε στο μέλλον, ίσως με την ευκαιρία του βραβείου Λούξ. Νομίζω καλό θα ήταν. Ε, ήθελα πάντα να πω ότι είσαι εξαιρετική και μου αρέσεις. Και δεν είμαι και ο μόνος. Θα μας λείψεις λοιπόν αυτό ήθελα να τονίσω. Σε ευχαριστώ πολύ Ντόρις. Καταρχήν Πολύ θα ήθελε ο Μάρκος Κούρια να είναι παρόν και να σου απευθύνει κάποιες, κάποια λέξεις, αλλά υποφέρει από πνευμονία, είναι ασθενής και για το λόγο αυτό δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα στη συνεδρίασή μας. Ευχόμαστε να επανέλθει η υγεία του στα φυσιολογικά της σύντομα. Η Doris Pack είναι μια πολύ γυναίκα έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά το μεγαλύτερο αυτό είναι η μεγάλη σκαρδιά. καρδιά όλοι μας ε, και εγώ φυσικά αισθανθήκαμε πάντα την παρουσίαση την παρουσία σου ότι πάντα μας ε, υπερασπίστηκες ε, ήμασταν σίγουροι για το έργο το οποίο έκανε η Επιτροπή μας. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία θετικά και πιστεύω ότι αυτό είναι σύμφω... με αυτό συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι και σας θυμόμαστε με ε, μεγάλη χαρά στα μελλοντικά χρόνια. Φυσικά θα μας λείψεις. Ο πιο έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, και εξ ονόματος της πολωνικής αντιπροσωπείας λείπουν μερικοί σήμερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά Δωρής θυμάμαι όταν πήγαμε στο Βρότσλαφ στην Πολωνία με την ευκαιρία μιας πολιτιστικής συνάντησης ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και έπρεπε τότε να αναλάβω την υποδοχή των Πολωνών Υπουργών και μου είπαν ότι ξέρουμε ότι η Δωρής ε, είναι χαρισματικό πρόσωπο και δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να την ε, διαχειριστείς. Τους είπα μην ανησυχείτε, είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά για όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί και τη συνεργασία μας και εγώ δεν θα κατεβώ στις εκλογές, αλλά θα με αντικαταστήσει ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Πολωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πακ, δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτήν την ειδονή να σας ευχαριστήσω. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών, νομίζω και οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε ε, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και για το φόρο τιμής που αποτίσατε στον Όμαρ Ταμπλίσκη. Θα μας λείψετε αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που το Προεδρείο σας ε, έδωσε τη θέση που αναφέρατε γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνέχεια για το βραβείο Λούξ. Λυπάμαι μόνο που δεν δίνεται μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το βραβείο που είναι μια μοναδική ευκαιρία να γίνουν συζητήσεις με τους συμπολίτε μας και μάλιστα σε όλες τις γλώσσες. Είναι πολύ μεγάλη η αξία του και συμβολική ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου σας ανέθεσε αυτό το καθήκον. Σας ευχαριστούμε πολύ. πρόεδρος της Οικων που αντικαθιστά την αίμα. Ναι, αντικαθιστώ την αίμα. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι παρόν εδώ για την τελευταία σου συνεδρίαση Δωρής και εγώ τη Δευτέρα έκανα την τελευταία μου συνεδρίαση. Θα ήθελα πρώτον εξ και της ΕΜΑΣ και των υπολείπων να σε ευχαριστήσω και εγώ για τον ηγετικό ρόλο που έπαιξε στην Επιτροπή μας. Εγώ πρωτοήρθα στο Κοινοβούλιο πριν από 15 χρόνια και θα μπορούσα να πω έτσι κάπως ευρύτερα ότι και στις διάσκεψεις των Προέδρων σε έχω δει και ήσουν πολύ στεναρή υπερασπίστρια προασπίστρια των δικαιωμάτων και δικαιοδοσιών του Κοινοβουλίου. Είμαι βέβαιος ότι και οι άλλοι συναδελφοί σου εδώ το ξέρουν και νομίζω ότι όταν έγινες πρόεδρος προς το τέλος της θητείας της διάσκεψης αυτής ε, έδειξες την αξία σου. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη, πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη χαρά που συνεργαστήκαμε μαζί σου. Βέβαια δεν ήμουν στην Επιτροπή αυτή, αλλά παρακολουθούσα τις εργασίες της, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα και νομίζω <coughs> ότι έκανες πολλά για να προωθήσεις τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ιδίως μέσω του βραβείου Λούξ. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να μπορέσει να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με την όθηση που της έδωσες. Σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά για όλα όσα έχεις κάνει, όχι μόνο στην Επιτροπή αυτή, αλλά και στο Κοινοβούλιο γενικότερα. Ξέχασα να ευχαριστήσω και όλους τους συμβούλους και το προσωπικό των ομάδων που εργάστηκαν και αυτοί τόσο καλά. Όχι μόνο από το ΕΛΚ που το γνωρίζω καλύτερα, αλλά και από τους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους, τους πράσινους της αριστεράς, καλά το είπα, καλά το είπα, τη αριστεράς και ε, είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Εδώ στην Επιτροπή ιδιαίτερα και με τους συναδέλφους και με το προσωπικό είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Εάν είναι κανείς από την Κομισιόν εδώ, τότε θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν. Α, ναι, εκεί είναι, εκεί είναι. Ευχαριστούμε πολύ και χαιρετίστε μου τους συναδέλφους σας. Στις 17 Μαρτίου κάναμε τον επίσημο αποχαιρετισμό. Δεν μην ξεχάσω και το τμήμα έρευνας που είναι εδώ μπροστά. Τώρα καθαρίζουν το γραφείο μου και βρίσκω διάφορα πράγματα που τα είχα ξεχάσει τα τελευταία χρόνια και μήνες και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά που κάνετε serious and to use it είναι πολύ καλή δουλειά και σε συνεργασία με εσά ετοιμάσαμε όλες μας τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να σας ξαναευχαριστήσω. Και τώρα λοιπόν κλείνουμε να ευχαριστήσω λοιπόν όλους και πάλι, να ευχαριστήσω και τους αναπληρωτές εδώ που αντικατέστησαν όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν εδώ σήμερα. Σας εύχομαι στους υποψήφιους τουλάχιστον έναν επιτυχή προεκλογικό αγώνα να επανεκλεγούν ανεξάρτητα από, το, την ομάδα στην οποία ε, εργάστηκαν και στην οποία ανήκουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Καλή επιτυχία και τώρα οριστικά και αμετάκλητα κλείνουμε.